Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της συνερήσιας διάταξης. Μηδέν-μηδέν είναι αν σας ενδιαφέρει ο αγώνας Γαλλία-Γερμανία. Το επόμενο θέμα είναι η χρησιμοποίηση παραδοσιακών ενδείξεων για κρασιά προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Mr. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η χρήση ορισμένων παραδοσιακών όρων για τα κρασιά είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ένωση. Μετά την μεταρρύθμιση των ίνων του 2008 δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο και κανόνες για την αναγνώριση, προστασία και χρήση τέτοιων παραδοσιακών ενειδίξεων. Καθόριζε ιδιαίτερα μία νέα διαδικασία για την προστασία των κρασιών που εφαρμοζόταν και σε ενωσιακούς ίνους και σε εξωενωσιακούς. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως πάντοτε έδειχναν κάποια αντίρρηση γιατί ως προς τη χρήση αυτών των παραδοσιακών ενδείξεων. Η Ινική Συμφωνία του 2006 Ένωσης ΕΠΑ ήταν η πρώτη συζήτηση για τη χρήση παραδοσιακών ενδείξεων για κρασιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ένωση και προέβλεπε ορισμένες εξαιρέσεις για τις εισαγωγές ίνων από τη ΣΥΠΑ που διέθεταν όμως trademark κατατεθειμένο στην Ένωση πριν από το Μάρτιο του 2006. Προβλέφτηκε και μία μεταβατική περίοδος τριών ετών ώστε τα κρασιά των ΙΠΑ που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακές ενδείξεις όπως σατό μέχρι να επιτραπεί η εμπορία τους. Η περίοδος αυτή έληξε τον Μάρτιο του 9. Τον Ιούνιο του 10 οι δύο κυριότερες ε, οργανώσεις, οι αμπελοϊνικές οργανώσεις των ΙΠΑ ζήτησαν την αναγνώριση της χρήσης του όρου ΣΑΤΟ στην Ένωση ως παραδοσιακού αμερικανικού όρου. Ο όρος λοιπόν ΣΑΤΟ χρησιμοποιείται εκτός από τη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο, στην Ιταλία, στη Χιλή και στον Καναδά. Ο όρος, ο ορισμός του υπάρχει αλλά δεν είναι ταυτόσιμο σε όλες αυτές τις χώρες. Αφού εξετάσαμε λοιπόν με βάση τη νέα διαδικασία, κάναμε μία δημοσίευση και η Γαλλία αντιτάχθηκε στην αναγνώριση αυτή λέγοντας ότι οι όροι των ΙΠΑ για τη χρήση του λέξης σατό θα οδηγούσαν τους Γάλλους καταναλωτές σε παραπλάνηση. Αυτό το γνωρίζουμε και ακόμη κάνουμε την αξιολόγηση. Θα χρειαστεί όσος χρόνος χρειαστεί. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπο, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, για δύο λεπτά, εξ ονόματος του ΕΛΚ, δίνω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Για άλλη μια φορά, θα πάρω το λόγο για να στηρίξω την κληρονομιά μας, την παράδοσή μας, την πολιτική μας κληρονομιά και την πνευματική μας κληρονομιά. Έναν τομέα στον οποίο η Ευρώπη συνεχίζει να είναι πρωταθλητής σαν παραγωγός, σαν εξαγωγός. Και πρόκειται για αυτή τη φορά να κατανοήσει η Επιτροπή ότι δεν μπορεί να υπάρχουν καταχρήσεις αιωνίως εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών κάποιων ενιών όπως σατό ή κλό για τα δικά τους κρασιά τα οποία εξάγουν και πολλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν για κάποιους λόγους εξωτερικής πολιτικής ή εμπορικούς λόγους να υποχωρήσουμε έτσι ώστε να αφήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες να καταχρώνται αυτές τις ενδείξεις και να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στην Ευρώπη κρασιά με την ονομασία Σατό ενώ δεν τηρούνται οι όροι. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην εφημερίδα των ε, κοινοτήτων δημοσιεύθηκε η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δήλωση της ε, ενάγουσας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι διέπουν έναν επαγγελματικό κλάδο ε, μιας τρίτης χώρας η οποία όμως δεν έχει συνοχή και δεν είναι και σοβαρή σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δυσάρεστη η αντικατάσταση του συναδέλφου εδώ. Είναι ένα θέμα τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Μπορείτε λοιπόν να του μεταβιβάσετε αυτό το μήνυμα και να του πείτε ποια είναι η άποψή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λούλινγκ. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επιτροπέ, συνάλφοι, η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη. Χρειάζεται να δείξουμε ευθύνη ε, σε ό,τι αφορά την προστασία της ενοπαραγωγής ε, μας της ελληνικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όλο και περισσότερα ε, φαινόμενα απομιμήσεων ε, βλέπουμε και η πρόταση αυτή για την αναγνώριση της χρήσης ενδείξεων όπως σατό και κλό από τις μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Μας εκπλήσει επίσης Κύριε Επίτροπε, αυτές είναι εμπορικές ε, πρακτικές που κατά, κατά πρώτον λόγο μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και κατά δεύτερο λόγο μπορούν να έχουν αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις ε, για του, τις ε, επιχειρήσεις που εμπορεύονται αυτά τα κρασιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι αμφισβητείται όλη η ευρωπαϊκή κληρονομιά ε, για παράδειγμα ε, προσέκο, ριόχα, σαμπάνια, απομιμήσεις αυτών εννοώ, ε, οι οποίες αμφισβητούν όλη την κατοχυρωμένη πολιτική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το κρασί, η εμπορική συμφωνία του 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ε, ανέστελε την άδεια χρήση ε, των όρων Σατό και Κλό το 2009, τρία χρόνια μετά δηλαδή, μετά από μια μεταβατική περίοδο. Ε, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την προστασία και την διαφάνεια των, ε, κατά, των ε, ενδείξεων στα κρασιά είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο προχωρημένη, η πιο πρωτοποριακή σε όλο τον κόσμο και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους παραπληροφόρηση, παραπλάνηση και απομιμήσεις. Παρ' όλα αυτά οι παραγωγοί ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν πλέον να παράγουν αυτά τα προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για όλα αυτά Βρισκόμαστε εδώ σήμερα προκειμένου να πείσουμε την ε, Κομισιόν ε, να μας ακούσει για να εγγυθούμε μια διαφανή αγορά με αμοιβαιότητα στις εμπορικές ε, πρακτικές. Είναι ασφαλώς σημαντικό να προωθήσουμε την διεθνή σύγκληση αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει με βάση τις δικούς μας κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό λεπτό, 1,5 λεπτό η κυρία Κρίσπεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μετά την πατάτα φλόρα, μετά τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς, μετά το ροζέ κρασί το οποίο φτιαχνόταν από κόκκινο και άσπρο κρασί αναμεμειγμένα. Σήμερα η Επιτροπή αναφέρεται στο θέμα αυτό που αφορά την χρήση του όρου σατό και κλό από Αμερικάνους παραγωγούς ίνου. Εγώ είμαι Γαλλίδα, αλλά δεν είναι μόνο γαλλικό το θέμα σήμερα. Υπάρχουν ε, παραγωγή κρασιού σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ακολουθούν μία μακρόχρονη παράδοση, πλούσια παράδοση, μία τεχνογνωσία. Και όσον αφορά παραδείγματο χάρη την λέξη «σατό» για την περιοχή του Μπορτό και «κλό» για τη Βουργουνδία, αυτοί οι όροι ανταποκρίνονται όχι μόνο σε ποιότητα, όχι μόνο σε παράδοση, αλλά και σε πολύ συγκεκριμένη πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι ένδειξεις αυτές που ακολουθούνται από συγκεκριμένες ε, ποιοτικές ε, ενδείξεις να συμπεριλαμβάνουν και μια συγκεκριμένη φήμη. Είναι σημαντικό λοιπόν κύριε Επίτροπε σήμερα να μην γίνεται καταχρηστική ε, ε, χρησιμοποίηση αυτών των όρων και να μην ε, υπάρχουν παραπλανητικές ενδείξεις που παραπλανούν και συγκεκριμένα τους καταναλωτές. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί παραγωγοί να χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο ε, όρους και ενδείξεις που σημαίνουν κάτι στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ. Μιλάμε για ένα θέμα που δημιουργεί πάθος, αλλά μην με υποχρεώσετε να σας ε, σταματήσω γιατί ξεπερνάτε το χρόνο σας. Κύριε Φερέιρα, ε, μετά την μεταρρύθμιση του ενοπαραγωγικού τομέα στην Πορτογαλία έχουμε μία ακόμα απειλή ε, σαν να μην έφτανε η δραματική κατάσταση στην κοιλάδα του Ντούρο ε, που, όπου ε, τα προκυπευτικά που παράγονται πολλούνται σε τιμές κάτω του κόστους τώρα βλέπουμε και την αμφισβήτηση ενδείξεων του κρασιού του Πόρτο που υπάρχουν εδώ και αιώνες παρά τις, ε, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ στις δικαστικές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τις ε, πόρτες στην ε, Αμερικανική εινοποιητική βιομηχανία για να επιβιώσει ως παράσιτο στην Ευρώπη. Μιλάμε για την ε, πιο ε, παλιά καθορισμένη περιοχή ε, εινοποίησης στον κόσμο η κοιλάδα του Ντούρο. θα πρέπει να αλλάξει στάση η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο για δύο λεπτά είναι ο κύριος Θέλω να συμπληρώσω την Astrid Luling που μίλησε πριν από λίγο που συνέκρινε τρει ορισμού, συγκρίνοντα τρει ορισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο όρο ΣΑΤΟ προστατεύεται. Σύμφωνα με τα άρθρα 118 ε, Β και Γ. Ε, το άρθρο 57 του 607-2009 δίνει ένα κοινοτικό ορισμό και ένα πλαίσιο εναρμονισμένης χρήσης ορισμένων παραδοσιακών ενδείξεων ε, που έχουν σχέση με την εινοπαραγωγή. Το 2007 και το 2009 η Κομισιόν, πριν τη συναπόφαση κύριε Επιτροπέ, η Κομισιόν έλεγε, λέω, ε, θεωρούσε ότι όλα αυτά ήταν λογικά. Ταυτόχρονα οι νομές Πολιτείες καθόρισαν στο ε, τίτλο 27.4.25 του κώδικά τους ε, την ε, ένδειξη σατό την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια ένας ομάδα παραγωγών για προϊόντα που προέρχονται από μούστο ως τμήμα της μάρκας ε, του εμπορικού σήματος. Πρόκειται λοιπόν για εμπορικό σήμα. Αυτός ο ορισμός προσπαθεί ε, να ε, μιμηθεί την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό ορισμό, αλλά δεν αντιστοιχεί σε αυτόν. Δεν αντιστοιχεί καν τον ε, ορισμό της Win America ε, η οποία ζήτησε τη χρήση του ορουσατό από τα μέλη του. Πιο αργά παρακαλώ τον Διακόπτη ο Πρόεδρος που, είναι, που αποτελεί διαφορετική, που ζητά μια διαφορε, ένα διαφορετικό ορισμό. Κανένα από τα στοιχεία της Επιτροπής ε, στη δημοσίευση στην ε, Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε, δεν ε, συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση της Wine America. Της Wine America. Ε, συνεπώς ε, η αίτηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά, κύριε Σαντρία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σήμερα νομίζω απαραίτητο κύριε Επίτροπέ μου η Κομισιόν να διασφαλίσει την απόλυτη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ετικέτες προέλευσης, για τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς ορισμούς γιατί η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται μόνο αν πληρούν τις ίδιες συνθήκες ή ανάλογες με εκείνες που απαιτούνται στα κράτη-μέλη. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε είναι παράνομο. Παράνομη αυτή η χρήση και δημιουργεί αθέμητο συνταγωνισμό μεταξύ Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών κρασιών που χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές ονομασίες Σατό και Κλό. Διότι τα Αμερικανικά κρασιά αντίθετα από τα Ευρωπαϊκά δεν τα επεξεργάζονται αποκλειστικά με βάση τον μούστο ούτε εινοποιούνται επιτόπου. Έπειτα αυτό αποτελεί παραπλάνηση του καταναλωτή και της καταναλώτριας διότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με συγκεκριμένο τόπο. Και έπειτα πρόκειται για παραπλάνηση και κατάχρηση της εργασίας πολλών δεκαετιών των παραγωγών μας. Άρα δεν έχουμε πια προστασία έναντι του παγκοσμίου ανταγωνισμού. Και αυτό μπορεί να αφορά και άλλα και άλλες παραδοσιακές ονομασίες, το Κάζα. Για την ευρωπαϊκή αμπελοεινοποιία λοιπόν κύριε Επίτροπε πρέπει να μας διασφαλίσετε ότι το αμερικανικό αίτημα είναι πράγματι αποδεκτό και απολύτως σύμφωνο με τους όρους που εφαρμόζονται και στην Ευρώπη και ιδίως τους ορισμούς που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Κύριε Δότα, πρέπει να σας πω ότι σας έκοψα μεν το λόγο, αλλά είναι ένα μηδέν υπέρ της Γαλλίας το μπάτσο. Signor Commissario, contro l'importazione da di prodotti contraffatti. Σιλβέστρης, ε, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν παρόμοια φαινόμενα απομιμήσεων και εισαγωγή του. Θέλω να σα παρουσιάσω μια πρόσφατη περίπτωση που εμφανίστηκε σε ε, όλα τα περιοδικά και τι εφημερίδες. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής κρασιού από χημικές, χημικής κατασκευής, παρασκευής σκόνες. Ε, υπάρχουν πολλά kit τα οποία πολλούνται και μπορούν να αγοραστούν μέσω ίντερνετ. Ε, ένα κουτί μέσα σε αυτό το κουτί υπάρχουν θειώδη και διάφορα άλλα ε, και διάφοροι μούστι για να δημιουργηθεί ζύμωση. Ε, Μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο kit και να φτιάξει το σπίτι κρασί με τέτοιου είδου χημικέ αειδίε και μάλιστα έρχονται αυτά τα kit μαζί και με μια ετικέτα ε, που ε, ε, έχει διάφορα αφημισμένα κρασιά εδώ κοιτάξτε το έχει μέχρι και μικρά σακουλάκια με ζάχαρη τα οποία, την οποία προσθέτουμε στα κίτ για να δημιουργηθεί αυτό το δίθεν κρασί λοιπόν υπάρχουν παραδοσιακές ενδείξεις στην Ευρώπη. Δεν μπορούν οι Πολιτείε να τι αντιγράφουν με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουν να τι χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να ακολουθούν τι αντίστοιχε πρακτικέ. Υπάρχουν ε, ονόματα όπω Κιάντι και Μαρσάλα, για παράδειγμα, τα οποία μιμούνται και ε, καταχρώνται οι Αμερικανοί. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχθούμε κάτι τέτοιο. Αυτά τα kit έχουν, είναι προϊόντα που, παράγονται στι ΗΠΑ. Αν αυτό είναι κρασί, τότε εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Για δύο λεπτά, η κυρία Χέρενς Καρσία έχει το λόγο. Παρόλη την Αμελονική ε, Συμφωνία του 2006 με, το, με τις ΗΠΑ, ε, στο πλαίσιο της οποίας κάναμε πολλές ε, παραχωρήσεις, οι ΗΠΑ δεν έκαναν καμία προσπάθεια κατά της κατάχρησης και της ιδιοποίησης των παραδοσιακών μας ενδείξεων. Μεταξύ αυτών και των ε, ονομασιών Χερέθ και Μάλαγα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει επιτέλους, να χρησιμοποιήσει τα μέσα, διπλωματικά μέσα που διαθέτει, έτσι ώστε οι ΗΠΑ να σταματήσουν με την παράνομη ε, χρήση αυτών των ονομασιών. Ε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόριου, μάλλον στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα μητρό παραδοσιακών ενδείξεων ε, και όταν οι Αμερικάνοι θέλουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδου ενδείξει, ε, τι θα κάνει η Κομισιόν, πώ θα εγγυηθεί ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί θα σέβονται τι ευρωπαϊκέ απαιτήσει Όταν η ίδια κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτει την ευρωπαϊκή πολιτική προστασία σε αυτών των ονομασιών. Επί τη ευκαιρία μεταξύ αυτών και η ονομασία σολέρα των κρασιών της Χερέθ. Ε, η Κομισιόν ε, θα προστατεύσει τα συμφέροντα των Αμερικανών ε, παραγωγών κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη χρήση παραδοσιακών ενδείξεων, ε, κάτι που θα αποτελέσει βέβαια ε, προηγούμενο στην αγορά. Η Κομισιόν με αυτόν τον ε, τρόπο υποσκάπτει την ευρωπαϊκή παραγωγή, η οποία πρέπει να σέβεται πολύ αυστηρού όρου ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των παραδοσιακών ενδείξεων. Πολύ περισσότερο που καταργούμε με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό ατού που έχουμε στο πλαίσιο μια συνολικότερη διαπραγμάτευση για την προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων στι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ. Ε, δεν είναι ο σωστό δρόμο αυτό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε του παραγωγού μα και την παραγωγή μα. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Ντόφμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρο, αξιότιμη κύριε Επίτροπο, συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να λειτουργήσουν οι εμπορικές συναλλαγές στον τομέα του κρασιού παγκοσμίω. Και θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι 23 εκατομμύρια λίτρα κρασιού εξάγονται και 13 εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η Αυτές οι εμπορικές συναλλαγές θα πρέπει να βασίζονται σε μια δίκαιη συναλλαγή, σε ένα δίκαιο σύστημα συναλλαγών και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι εμπεριέχει αυτό το προϊόν που αγοράζει και ονομάζεται κρασί. Οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτό που τους ζητείτε βάσει αυτών των δίκαιων εμπορικών συναλλαγών. Όταν παραδείγματο χάρη πολλούν ένα προϊόν σαν προσέκο, σαν σαμπάνια ή σαν κρασί, αυτό το προϊόν να είναι πραγματικά προσέκο κρασί. Όπως ξέρετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε παράγουν πολλά εκατομμύρια λίτρα κρασιού, από τα οποία εξάγουν ένα σημαντικό αριθμό, εισάγουν όμως πολύ περισσότερο ε, κρασί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι ε, εξάγουν σε εμά. Έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον να συνεχίσουν να λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Νόμαν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, οποιαδήποτε χρήση παραδοσιακών ενδείξεων όπως οι λέξεις vintage των κρασιών του Πορτό ε, και άλλες ε, αποτελεί ε, απειλή και επίθεση εναντίον των παραγωγών και της παραγωγής μας. Πρόκειται για απειλή απέναντι και στους κατανοητέ διότι τους παραπλανούν αυτές οι ενδείξεις. Πρόκειται επίσης ε, για επιθέσεις εναντίον των παραγωγών διότι ιδιοποιούνται την δουλειά τους ε, ε, και τους αφαιρούν πόρους ε, τα, τους οποίους ε, έχουν ε, δημιουργήσει μετά από δουλειά πολλών πολλών χρόνων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμφέροντα των καταναλωτών και ταυτόχρονα να ακολουθήσουμε μια πολιτική προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων Ήδη δόθηκαν τρία χρόνια παράτασης ε, περίοδου ε, και αυτό δεν μείωσε τις ε, παραβάσεις. Ελπίζαμε ότι αυτή η παράταση θα βοηθούσε στην παρεμπόδιση ε, παραβάσεων που έγιναν εκτός, γινόντουσαν εκτός συμφωνίας. Δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο. Δημιουργήθηκε μάλιστα και προηγούμενο, που δεν είναι δυνατόν να το διαιωνίσουμε. Το πρόβλημα δεν υφίσταται μόνο με τις ΗΠΑ. Ε, υπάρχει μια απειλή γενικότερα από την Αμερική και από, από άλλες τρίτες ε, χώρες που θέλουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ονομασίες όπως για παράδειγμα η Κίνα, γιατί η Κίνα μπορεί να προτιμήσει να εισάγει τέτοιου κρασιά με τέτοιες ονομασίες από τι ΗΠΑ αντί από την Ευρώπη. Συνεπώ, ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να κλείσει οριστικά και να ληφθούν αυστηρά μέτρα έναντι τη ιδιοποίηση των ενδείξεών μας και των απομιμήσεων. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, η κυρία Κάστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν αναφερόμαστε σε ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης για το κρασί, σαφώς δημιουργούνται τέτοιες έντονες συζητήσεις. Ξέρουμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την παραγωγή, ενώ η ε, ο Αμερικανικό κλάδο των ινοπαραγωγών έχει μια τελείως διαφορετική στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι για μας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, γιατί ήδη από το 2006 έχουμε μια συμφωνία που έχει τεθεί σε ισχύ για τον τομέα αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λύση όμως δεν βρέθηκε και τα προβλήματα συνεχίζουν. Βλέπουμε ότι Υπάρχουν κάποιες γενικές ονομασίες κρασιών και όταν δεν περιέχονται παροδοσιακές ενδείξεις, τα αμερικανικά προϊόντα δεν δημιουργούν πρόβλημα. Όμως το θέμα που συζητούμε σήμερα δεν έχει λυθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναζητήσω στην Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι το πρότυπο που προσπαθούμε εδώ να δημιουργήσουμε θα πρέπει να εφαρμοστεί στον τομέα του κρασιού και από μέρους της Επιτροπής θα περίμενα κάτι πιο συγκεκριμένο και να μας εξηγήσει με ποιο τρόπο θεωρεί ότι μπορεί να προστατεύσει τους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και τους Ευρωπαίους παραγωγούς καθώς και τους αντίστοιχους Αμερικάνους. Πώς μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες εγγύησεις. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Κλάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ευαίσθητο, αν θέλετε, προϊόν το κρασί, γιατί είναι την ίδια ώρα κάτι το οποίο μας θυμίζει την πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν και η λύση του προβλήματος που συζητούμε σήμερα μας θέτει διάφορες πολύ σημαντικές προκλήσεις. Είναι απαραίτητο σήμερα να δούμε ποιες είναι αυτές οι παραδοσιακές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η λέξη σατό, η λέξη κλό σημαίνει κάτι για τους Γάλλους, για τους ε, Λουξεμβούριους. Είναι κάτι που για έναν Γερμανό παραδείγματος χάριν δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Σημαίνει παραδείγματος χάριν ότι όλα τα σταφύλια, όλα τα αμπέλια ανήκουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και πολλές φορές σε καμία συγκεκριμένη πολύ μικρή περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικό διότι σημαίνει κάτι για την προέλευση αυτού του κρασιού. Σημαίνει κάτι για τον τρόπο παραγωγής αυτού του προϊόντος. Το θέμα δεν είναι αν είναι καλό ή κακό, αν θέλετε, το κρασί. Η γερμανική γλώσσα, παραδείγματος χάρη, δεν περιέχει τόσες πολλές ε, λεπτομέρειες για την περιγραφή αυτού του προϊόντος. Η σαμπάνια, το άσπρο κρασί, όλα αυτά τα προϊόντα έχουν τη θέση τους στην αγορά με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το γερμανικό σεκτ επίσης έχει βρει τη θέση του στην αγορά. Είναι λοιπόν σημαντικό οι χώρες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα αλλά έχουν παρόλα αυτά δεχτεί αυτές τις ενδείξεις να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο πίσω από αυτούς τους όρους και όλα αυτά ρυθμίζονται νομικά. Και για μας κύριε Επίτροπε όλα αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Σάντσες Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2012 ήδη είχαμε ανησυχήσει για την πρόταση της Κομισιόν να επιτρέψει την πώληση στην Ένωση Αμερικανικών κρασιών που να αναφέρουν την ένδειξη σατό και κλό που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη Γαλλία για να εγγυηθούν στον καταναλωτή και την καταναλώτρια την ποιότητα του προϊόντος. Η χρήση τέτοιων όρων σημαίνει κανονικά ότι προέρχεται από έλεγχο της προέλευσης με πολύ συγκεκριμένους όρους. Ενώ τα αμερικανικά κρασιά δεν έχουν καμία εγγύηση προέλευσης και είναι καθαρά βιομηχανικής παρασκευής εφόσον θέλουμε ποιοτική ε, παραγωγή κρασιών πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πρόκειται για τρομερή κατάχρηση και παραπλάνηση. Ελπίζω η Κομισιόν να έλθει στα σύγκαλά της και να μετανιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Mr. President, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους για την συνεισφορά σας. Σημείωσα προσεκτικά τις ανησυχίες σας και θα τις θέσω υπόψη του συναδέλφου του κυρίου Τσιόλος, που είναι υπεύθυνο για το ζήτημα. Ε, σύμφωνα και με τα όσα ζήτησε η κυρία Λούλινγκ. Θα επαναλάβω αυτά που είπα και στην αρχική μου εισαγωγή. Η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά την ευαισθησία ε, το, του θέματος, το ευαίσθητο του θέματος και τις πολιτικές του προεκτάσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Σχετικά με, τις, ε, με τα αιτήματα των ΗΠΑ, η νική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τύχει σεβασμού και από τις δύο πλευρές. Ε, πτήσεις των ΗΠΑ υπευλήθηκαν σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις γεωγραφικές ενδείξεις μας. Ε, όμως, παραδοσιακοί όροι δεν αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, αποτελούν τμήματα της επισήμανσης των προϊόντων. Τούτου λεχθέντος η Κομισιόν εξακολουθεί να μελετά τις, ε, τα αιτήματα. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Συνεχίζουμε την εξέταση αυτών των αιτημάτων και σίγουρα θα λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα των ε, παραγωγών ίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εδώ λοιπόν αφού μιλήσαμε και για τα κρασιά ελπίζω να μπορέσετε να πιείτε και ένα ποτήρι. Λίγη συνεδρίαση εδώ. Θα επαναληφθεί αύριο το πρωί και υπάρχει η περίσσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και τους κυρίους ε, κλητήρες και τους διερμηνείς και διερμηνεύτριες.